Okay. Uh, welcome everybody. I will speak in Swedish for the first minutes and then we on during the... θα, ξεκινήσω, θα μιλήσω σουηδικά για τα πρώτα λεπτά και στη συνέχεια θα αλλάξουμε στα αγγλικά. Θα μιλήσω αγγλικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτή την συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης και ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε λίγο, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Η συνεδρίαση των συντονιστών είναι το πρώτο σημείο στην ημερησία διάταξη. Το ολοκληρώσαμε και όπως ε, λέω συνήθως ε, μπορείτε να μιλάτε όπου θέλετε εκτός από αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, το δεύτερο σημείο είναι η έγκριση της ημερησίας διάταξης. Κανείς δεν έχει ζητήσει κάποιες τροποποιήσεις. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι εγκρίνεται. Σημείο 3, ανακοινώσει του Προέδρου. Και όπως θα ξέρετε, η κυρία Μπέργμαν ε, την καλωσορίζουμε και θέλουμε να καλωσορίσουμε και την κυρία Κριστίνα Μορβάη από τους μη εγγεγραμμένους, μια συνάδελφος. Και να πω ότι η κυρία Μάης δεν είναι πλέον ε, μετακτικό τακτικό μέλος στην ομάδα αυτή και να σας πω ότι στις 9 Οκτωβρίου είχα μία κοινή συνεδρίαση και στην αίθουσα θα βρείτε ένα χρονοδιάγραμμα με τη συνεδρία της Επιτροπής μας ε, το 2013. Έχει μοιραστεί το έγγραφο αυτό. Λοιπόν, Περνάμε στο σημείο 4, ανακοινώσει του Πρόεδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. Έχουμε μοιράσει τις συστάσεις αυτές, δεν έχουμε λάβει κάποιες αντιρρήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνονται και μπορούμε να τις προσθέσουμε στα πρακτικά. Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω μία μικρή αλλαγή στο πρωτόκολλο της 25 ε, Σεπτεμβρίου 2011. Πρόκειται να κάνουμε μια προσαρμογή εκεί και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ηλεκτρονική μας ψηφοφορία. Okay, then we start the voting. Uh, Ξεκινάνε οι ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με το, τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία ορίζον 2020 και θέλω να ρωτήσω εάν ο εισηγητής, η εισηγήτρια θέλει τον λόγο η κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν με ε, τροπολογίες διότι θέλουμε τα προβλέματά μας να περιληφθούν στον ορίζοντα 2020 η αριστεία, οι αλλαγές στην κοινωνία καθώς και η βασική έρευνα και η ανθρώπινη πόροι θα ασχοληθούμε και με την ε, κατανομή των πόρων κατά τρόπον ώστε οι ερευνητές άντρες και γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες ε, εκτελέσεως ερεύνης και να έχουν την δυνατότητα για ε, επαγγελματική πρόθεση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε για να προωθηθούμε και ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ψήφιση αυτής της γνωμοδοτήσεως. Ευχαριστώ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ε, κυρία Κορνέλησεν, βλέπω ότι είσαστε έτοιμοι να ψηφίσετε ε, και ξεκινάμε με την τροπολογία 30. Τροπολογία 30. Ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά έχουμε την τροπολογία 33 σε δύο τμήματα ψηφίζουμε καταρχήν το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι χρειάζεται ε, έλεγχος και ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. And the vote is closed. Έληξε. Απερίφθη. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω και εδώ χρειάζεται έλεγχος. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 8. Λίγη. Εγκρίθηκε νομίζω. Με συγχωρείτε, δεν τα είχα δει, δει καλά εγώ. Ε, τροπολογία 34, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Έλεγχος στην 35. Έλεγχος ηλεκτρονικός ξεκινά. Έληξε. Ενεκρίθη. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 37 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 38 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 39 υπέρ κατά αποχές Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έληξε. Ενεκρίθη. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη δηλαδή καταπίπτει 23 και ούτω καθεξής και πάμε στις 49 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 50 με μία ε, προφορική ψηφοφορία, ε, τροπολογία, οπότε αν δεν έχετε ε, αντίρρηση, τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν πολύ σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην τροπολογία 53 ξεκινά. Έληξε, ενεκρίθη. Είναι πολύ σαφές. Αλλά τουλάχιστον δεν ήταν πολύ προφανές, ίσως γιατί δεν ήταν αρκετά ψηλά τα χέρια αν κάποιος δεν ψηφίζει δεν είμαι σε θέση να το αντιληφθώ. 54 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος στην τροπολογία 54. Ηλεκτρονικά. Ξεκινά. Λίγη ενεκρίθη 55 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 56 είναι χωριστή ε, ψηφοφορία ψηφίζουμε το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά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 Είμαι σίγουρος ότι είδα ένα σωρό χέρια όταν είχα ε, ζητήσει ποιος είναι κατά. Ίσως είναι η καθυστέρηση της μετάφρασης, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 65, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 και 67 είναι ταυτόσιμες. Τις ψηφίζουμε μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 και 70 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 και 77 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 78 και 79 επίσης ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 80 και 81 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 82 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθησαν 83 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 84 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. 88 υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. 89 υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. 90 υπέρ, με συγχωρείτε, 89 και 90 είναι ταυτόσιμες, οπότε προχωράμε στην 91. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 95 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος στην 95. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 95 ηλεκτρονικά. Πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 τι είπατε? Εκτός μικροφώνου διάλογος. Τι εννοείται λέει ο πρόεδρος. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέτε, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε την 127. Υπέρ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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το ψήφισμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάει τώρα πέρας και εγκρίνεται σαφώς ευχαριστώ λοιπόν ε, την εισηγήτρια. On to, uh, να περάσουμε στο σημείο 7, κατάρτιση του προγράμματος δικαιώματα και ηθαδένεια για την περίοδο 2014-2020. Η συγκεκριτή θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Απλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν ε, τροπολογίες ε, και ε, τους συναδέλφους εισηγητές και εισηγήτριες που ουσιαστικά με τις τροπολογίες τους έκαναν πιο συνεκτικό και πιο απλό το κείμενο και όλες οι τροπολογίες ήταν προς την διακατεύθυνση, δηλαδή να δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα αυτή την περίοδο 2014-2020 και θα ε, συμπεριληφθεί το πρόγραμμα Δάφνη στο πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια. Επίσης, ενισχύονται οι στόχοι καταπολέμησης της βίας κατά των νέων των παιδιών και των γυναικών και τέλος ε, Θέλουμε να μην μειωθεί η χρηματοδότηση, τα κονδύλια για το πρόγραμμα αυτό. Και μάλιστα θα θέλαμε και περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ λοιπόν όλους και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας πω το εξής. Τουλάχιστον στη δική μου σελίδα υπαριθμών 6 το εκτιμώντας 6, τροπολογία 3, λέει στη δεξιά κολόνα ότι καταπίπτει αν υιοθετηθεί η τροπολογία 25. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή θα πρέπει να συνδυαστεί με την τροπολογία 25. Έτσι λοιπόν όταν θα φτάσουμε στην τροπολογία 3 θα το συζητήσουμε. Θα Τουλάχιστον να σα το γνωστοποιήσω. Ξεκινάμε τώρα την ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 51 υπέρ. Παρακαλώ, με ένα χειρό. κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Δηλαδή καταπληκτή 52. Περνάμε στην τροπολογία 9 υπέρ. Κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει 55 55, 54, 56 καταπίπτουν και αποσύρεται 57. Περνάμε στην τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε. Για την τροπολογία 58 άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 58. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 2. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Γκρίνεται. Επομένω, όλε τι τροπολογίε καταπληκτούν. Πάμε λοιπόν στο συμβιβασμό υπερθμό 3. Υπέρ, κατά, ποιε, Γκρίνεται. Επίση, καταπληκτούν και άλλε τοπολογίε. Πάμε λοιπόν στην 63. Υπέρ, κατά, ποιε, Γκρίνεται. Τοπολογία 66. Υπέρ, κατά, ποιε, εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε νομίζω την 71 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 73 υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός περιθμών 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Συγγνώμη. 82 Ψηφίζουμε την τροπολογία 82 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβέσμος περιθμών 5 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Και αυτό σημαίνει ότι πολλές τροπολογίες καταπίπτουν, επομένως περνάμε στην 88 τροπολογία υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία υπαρθμών 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 αποσύρεται. Και έχουμε την τροπολογία 96 που είναι τμήματική ψηφοφορία. Περνάμε με το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πρέπει να περάσουμε στην τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Να περάσουμε λοιπόν στην τροπολογία περιθμών 99, υπέρ παρακαλώ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Μάλλον να ελέγξουμε την 99, λέει ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 99. Πέρας. Απορρίπτεται, λίγο, ο πρόεδρος. 100 περ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ είναι προφορική τροπολογία υπάρχει αντίρρηση από κάποιο συνάδελφο όχι Κάποιος πρέπει να παρουσιάσει αυτή την τροπολογία. Παρακαλώ κυρία Κώστα. Η τροπολογία Childers ουσιαστικά λέει ότι η έκθεση επί του ετησίου προγράμματος πρέπει να βασίζεται σε δύο συγκεκριμένα άρθρα που είναι οι στόχοι. Η δική μας τροπολογία προβλέπει να αναφερόμαστε ιδίω σε αυτά τα δύο άρθρα, όχι μόνο σε αυτά τα δύο άρθρα. Το in particular δηλαδή θέλουμε να βάλουμε εδώ. Αυτή είναι η τροπολογία. Να μην έχουμε μόνο αυτά τα δύο άρθρα. Το in particular θέλουμε να προσθέσουμε, μάλιστα. Ακριβώς, λέει ο Πρόεδρος, αντιρρήσεις. Όχι. Να ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 101 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, εποχές, νομίζω απορρίπτεται να ελέγξουμε την 103. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 103. Πέντε λείπουν, λέει ο πρόεδρος, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 104, υπέρ. Κατά. Εποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν σηκώνουν όλοι τα χέρια τους. Και... Αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας, ε, είναι δύσκολο για μένα ως πρόεδρο να δω. Να ελέγξουμε την 104. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Νομίζω τρεις είχαν σηκώσει το χέρι του υπέρ και δύο κατά. Οι υπόλοιποι 27... Σχόλιο εκτό μικροφώνου. Δεν θα απαντήσω, λέει ο πρόεδρο. Περνάμε στην τροπολογία 105. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι καταπληκτική η τροπολογία παρθμών 21. Περνάμε λοιπόν στην 23. Τμηματική ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. η δύο λοιπόν καταπίπτει. Περνάμε στην 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ Κατά. Όχι. Είπα ότι θα ψηφίσουμε επί της 3. Δεν καταπίπτει γιατί είναι λάθος αυτό που λέει στο έγγραφο. Λοιπόν, τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Σας παρακαλώ. 26 καταπίπτει και περνάμε στην 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 29. Κοιτάξτε, και πάλι είχα 4 υπέρ, 5 κατά. Θέλω να δω και του συντονιστέ, αλλά ούτε αυτού του βλέπω το ψηφίσουν. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, έρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 29. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Και άλλη προφορική τροπολογία, ούτε εδώ υπάρχει αντίρρηση. Ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός περιθμών 1 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι πολλές τροπολογίες καταπίπτουν. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην υπαριθμόν 35 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την υπαριθμόν 35, έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Θυματική ψηφορία για την 36. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Οχέ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Να ελέγξουμε. Το πρώτο τμήμα για την τροπολογία 36. Κατόπιν περνάμε στο δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. πίπτη 37, περνάμε στην 38, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Και είναι το με την 39. Περνάμε λοιπόν στην υπερθυμόν 40, υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. 41 τμήματική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ. Συγγνώμη, αποσύρεται, αποσύρεται αυτή. Και καταπέπτει 43, επομένω πάμε στην 6. Τροπολογία παριθμών 6. Υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά εποχές Γκρίνεται. 49. 49 και 50 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. πιπτή 8. Περνάμε στη 19. Υπέρ. Κατά. Εποχές γκρίνεται. Και τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία το σύνολο του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται, από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Πάμε στο 8ο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για συντονισμό οικονομικής πολιτικής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 Έλεγχος της 17. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τροπολογία 17. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω... Ας ελέγξουμε την τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ έλεγχος για την 21. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 21.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 Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για την 32. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν ένας τροπολογής και φτάνουν στην τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα, το ίδιο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάει τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Τώρα προχωράμε στο 9 την ενδιάμεση έκθεση εν ώψη της θετικής έκβασης της διαδικασίας έγκρισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Αφού η συγγήτρια δεν θέλει τον λόγο, ξεκινάμε με τη ψηφοφορία, τροπολογία 2 απορρίπτεται, ε, τροπολογία 3 υιοθετήθηκε, 4 υπέρ, κατά. Ποιος είναι υπέρ της τέσσερα. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Υιοθετήθηκε. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα 6 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 8 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 10 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 13 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 14 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 16 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ένα υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. Τώρα ψηφίζουμε ολόκληρο το ψήφισμα ηλεκτρονικά. Ξεκινάμε. Λίγοι ενεκρίθη. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Προχωράμε στο 10 πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μήπως η, εισηγήτρια θέλει το λόγο, η κυρία Γιανακουδάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας πω σχετικά με την συμβιβαστική ένα ότι έχουμε μία τεχνική τροπολογία και χρειάστηκε να αλλάξουμε ε, τη διατύπωση flexible training διότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να προβεί σε ε, εκπαίδευση αλλά ε, καθοδήγηση για για εκπαίδευση, δηλαδή να προωθήσουμε την εκπαίδευση χωρίς όμως ουσιαστικά να την προσφέρουμε. Ο ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Ξεκινάμε με την τροπολογία 35. Υπέρ, κατά, αποχές, απο, ε, ε, απορρίπτεται. 36. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, κρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 39 καταπίπτει ψηφίζουμε τη 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 41 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 42 υπέρ κατά αποχές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 απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος για, τις, για τη 10. Ξεκινάει. Λίγη. Απερίφθη. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ε, ψηφίζουμε την τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απερίφθη 12 ε, υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 58 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την 58 και ξεκινάμε ηλεκτρονικό έλεγχο της 58. Έληξε. Ενεκρίθη. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ηλεκτρονικός έλεγχος στις 14 ξεκινά λίγη ενεκρίθη πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το 60 καταπίπτει ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 17 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη Ας ελέγξουμε την 17 ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. Ενεκρίθη. Οπότε το 15 καταργείται και τώρα ψηφίζουμε την 16. Μάλλον την 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 3 ε, υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 21 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 22 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 23 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 27 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 28 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 29 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 30 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 4 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 5 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 6 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 31 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη Συμβιβαστική 1. Και αυτή είναι μία προφορική τροπολογία. Έχετε αντιρρήσεις. Όχι, τότε ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και προχωράμε στην 33. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε όλο το ψήφισμα ηλεκτρονικά ξεκινά η ψηφοφορία Λίγοι και σαφώς ενεκρίθηκε ευχαριστώ την εισηγήτρια meest. Yeah, exactly. Uh, then going on to the next, and that's uh, uh, item 11, Creative Europe Program. περάσουμε στο επόμενο σημείο, πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Έχουμε δύο προφορικές τροπολογίες. Να σας ρωτήσω αν ε, υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτές τις προφορικές τροπολογίες. Μπορούμε λοιπόν να τις ψηφίσουμε ομαδικά. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο πλέον να σας πω ότι η Επιτροπή από την Επιτροπή Πολιτισμού για τη το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και λέω τώρα ότι εγώ συμφωνώ με την ουσία αυτών των τροπολογιών αλλά ήθελα να καθησυχάσω εδώ τη συναδέλφους από την Επιτροπή ότι στο δικό μου κείμενο έχω βάλει κάτι συγκεκριμένο σημείο στο διατακτικό για να υποστηρίξω κυρίως ε, τα έργα των ε, γυναικών ε, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 12, αναθεώρηση τη στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε έτοιμα για τη μηματική ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη τροπολογία. μόνο 1. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο, 13 αποφάσεις στον τομέα των περιουσιακών ε, σχέσεων των καταχωρημένων συντρόφων. Θέλει η συγκήτρια το λόγο. Όχι, ωραία, να περάσουμε στην ψηφοφορία για όλες αυτές τις τροπολογίες. Ξεκινάμε με την υπαριθμό 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εποχές νομίζω απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος αλλά να ελέγξουμε την υπαριθμόν 5 για να είμαστε σίγουροι άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Thank you very much for the votes. Σας ευχαριστώ για τις ψηφοφορίες και τώρα θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια και θα μιλήσω σου ειδικά. Eh, eh, Ωραία. Να συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μα Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και υπάρχουν αρκετά που μπορούμε να συζητήσουμε επί του θέματος αυτού και είναι ιδιαίτερα και, επί, και ιδιαίτερα επίκαιρο. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στην κυρία Κράτσα.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 ε, προετοιμάζει την υποβολή μιας πρότασης όπου δεν ξέρουμε την τελική της μορφή αλλά υποθέτουμε ότι η πρόταση αυτή ε, έχει να κάνει με υποχρεωτική ποσόστοση στα συμβούλια ε, τα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι είναι ένα, μια ευτυχής κατάληξη της πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου μας και της Επιτροπής μας να ανοίξουμε τον διάλογο δημόσια για το θέμα αυτό και να έχουμε μια πρόταση της Επιτροπής. Ε, στι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να προκαταβάλουν ε, την ε, ε, πρωτοβουλία της Επιτροπής, κάτι που δεν είναι σωστό διότι παρακάμπτεται έτσι η, η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θα πρέπει η Επιτροπή να κάνει την πρότασή της, να την εξετάσουμε εμείς και το Συμβούλιο και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Ε, ξέρουμε ότι η Ευρώπη κτίζεται σε δύο επίπεδα, εθνικό και ευρωπαϊκό. Δεν, ε, αφήνουμε, δεν είμαστε αδιάφοροι για, το, για την άποψη και τον ρόλο των κυβερνήσεων, αλλά τουλάχιστον πρέπει να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή διαδικασία. Δηλαδή το λέω αυτό ανεξάρτητα της ουσίας, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε ενοχλημένοι, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ενοχλημένοι, από αυτή την διαστρέβλωση της διαδικασίας της νομοθετικής που επιχειρείται από τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, επί της ουσίας, νομίζω ότι ε, ε, ε, είναι ευτυχής κατάληξη, επαναλαμβάνω, και εμείς πρέπει να σταθούμε προσεκτικά και θετικά σε αυτή την πρόταση της Επιτροπής. όταν θα έρθει η πρόταση θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις τροπολογίες μας και την επεξεργασία μας. Αλλά ε, πιστεύω ότι την στιγμή αυτή όπου υπάρχει αυτή η, η ατμόσφαιρα ότι υπάρχει μια μειοψηφία μπλοκαρίσματος ήδη της πρωτοβουλίας επιτροπής νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να αντιδράσουμε ε, θυμίζοντας το ευρωπαϊκό συμφέρον, την ευρωπαϊκή διαδικασία, την ομοθετική και ενθαρρύνοντας και τις κυβερνήσεις μας και τους ε, και τα μέλη της Επιτροπής να έχουν μια θετική ε, προσέγγιση του θέματος αυτού. Και πιστεύω ότι ε, θεωρώ απαράδεκτο αυτό το, το κλίμα το, το αρνητικό και το καχύποπτο που έχει δημιουργηθεί πίσω, ε, γύρω από αυτή την πρωτοβουλία, την ανακοίνωση δηλαδή, της κυρίας Ρέντιγκορ θα υποβάλει την πρωτοβουλία, διότι την εποχή αυτή της κρίσης, όπου σίγουρα η Ευρώπη βάλεται και ουσιαστικά και σημειολογικά ουσιαστικά διότι δεν μπορεί να δώσει, να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης που είναι απαραίτητοι για την ευημερία της και την ανταγωνιστικότητά της, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή, που δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα α, των νέων ανθρώπων που πλήττονται ιδιαίτερα από την, ε, από την ε, ενεργία, να δώσει ε, δυνατότητες στις επιχειρήσεις μας να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, να είναι ανταγωνιστικές στον κόσμο, ε, πολλές φορές αισθανόμαστε προσεκτικά στις απαιτήσει μας όταν έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος. γιατί ξέρουμε τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Αλλά για κάτι το οποίο δεν έχει κανένα κόστος. Αντίθετα, έχουμε όλες τις μελέτες από την Ευρώπη, από την Αμερική, από άλλες αναπτυγμένες ε, οικονομίες, από ερευνητικά κέντρα, ότι θα συμβάλλει μια τέτοια μέθοδος στη δραστηριοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ε, ε, συμμετοχή ταλέντων μέσα στην οικονομική διαδικασία θα δώσει άλλες ε, ε, επιδόσεις και, και βιωσιμότητα επιχειρήσεις, είναι κρίμα να είμαστε έτσι μεμψίμυροι. Νομίζω ότι το θέμα πρέπει να ξεφύγει από και τα ιδεολογικά πλαίσια και τα παραδοσιακά ε, στερεότυπα. Πρέπει να δούμε μπροστά για την κοινωνία και την οικονομία. Και νομίζω ότι πρέπει εμείς να κάνουμε σαφές, σαφές το μήνυμα αυτό ήδη προτού μας έλθει η πρόταση η νομοθετική. Διότι αν μείνουμε αδρανείς, από ό,τι φαίνεται μπορεί να μην μας έρθει η πρόταση. Εδώ είμαστε μπροστά σε δύο δρόμους. Το, το βλέπω στην κοινή γνώμη με την οποία επικοινωνώ. Πιστεύω ότι και εσείς θα διαπιστώνετε το ίδιο. Απ' τη μια μεριά υπάρχει αίσθηση ότι τώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα, κρίση δημοσιονομική, ε, ε, σωτηρία του ευρώ, διασφάλιση των αρνητικών επιπτώσεων, αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που έχει η κρίση στην Ευρωζώνη στις χώρες εκτός Ευρωζώνης και πολλοί λένε δεν είναι τώρα η ώρα να συζητήσουμε αυτό το θέμα, δεν έχει θέση μέσα στα προβλήματα και τις προτεραιότητες της Ευρώπης. Αντίθετα, εμείς πρέπει να σταθούμε, ε, να υψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε ότι μια Ευρώπη όπως την επιθυμούμε δεν χτίζεται μόνο διάστατα, μόνο με την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Υπάρχουν ε, πληθώρα ε, θεμάτων τα οποία είναι καθημερινή μας ενασχόληση και δεύτερον, και αν σταθούμε στην προτεραιότητα της κρίσης, επαναλαμβάνω οι μελέτες μας λένε ότι η εμπλοκή των γυναικών στη διοίκηση των επιχειρήσεων θα βοηθήσει την Ευρώπη και στην ανάκαμψη και στην αντιμετώπιση της κρίσης. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώρια να μένουμε αδρανείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τους συντονιστές καταρχήν. Κυρία Κορνέλησον, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κράτσα για την εισαγωγική σας. Όλοι έχουμε διαβάσει το σχέδιο κειμένου. Δεν είναι βεβαίω επίσημο ακόμη το κείμενο. Έχει διαρρεύσει, αλλά χαίρομαι που υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο χαρτί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στην κυρία Ρέντινγκ, να δείξουμε υποστήριξη και από όσε πλευρές είναι δυνατόν να τις δείξουμε ότι πράγματι θα έπρεπε να προωθήσει το ζήτημα αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Κράτσα ότι ουσιαστικά το Συμβούλιο μας προσβάλλει καθώς δεν αφήνει τη δημοκρατική διαδικασία να ακολουθήσει την οδό της και πραγματικά προσβάλλει και τον εαυτό του. Όχι όλο το Συμβούλιο, αλλά κάποιες χώρες. Καθώς δεν θέλουν μία ανοιχτή και δημόσια συζήτηση. Τελικά, όταν ε, θα έλθει επιτάπητος ε, θα έχουμε μια συζήτηση και θα πούν ε, όχι δεν το θέλουμε αυτό και έχουμε ουσιαστικά τον αριθμό να τον μπλοκάρουμε. Όμως καθώς δεν έχει συζητηθεί ακόμη είναι πραγματικά ντροπιαστικό για αυτούς να φοβούνται την δημόσια συζήτηση. Αν, αν εξαρτώταν από μένα, εγώ θα ζητούσα από τον πρόεδρο της Επιτροπής από την ίδια την Επιτροπή να γράψει μια επιστολή προς την κυρία Ρέντινγκ και να την υποστηρίξει. Και ουσιαστικά, αν δεν υπάρχει συνένεση, τουλάχιστον ε, μια συμμαχία των προθήμων από αυτήν την Επιτροπή θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Μάλιστα, σας ευχαριστώ για την πρόταση αυτή. Τόμψεν, δεύτερη συγγήτρια. Εγώ ανησυχώ για την ε, διαδικασία και χάρηκα πάρα πολύ με όσα είπε η κυρία Κράτσα για το πώς πρέπει εμείς να το χειριστούμε από τη δική μας πλευρά, από το Κοινοβούλιο. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί αυτό αποτελεί συνέπεια της συνθήκης της Λισαβόνας. Το Συμβούλιο δεν είναι έτοιμο το Κοινοβούλιο να επηρεάσει επίσης. Το είδαμε αυτό και κατά τη διάρκεια της Προεδρία της Δανίας ε, με την υπόθεση Σέγγεν, όπου το Συμβούλιο αποφάσισε χωρίς να λάβει υπόψη την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πάλι αυτό βλέπουμε εδώ, αλλά αυτή τη φορά είναι ακόμη χειρότερο, καθώς ε, μπλοκάρουν μια οδηγία πριν να έχει καν παρουσιαστεί. Και νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε το καλό παράδειγμα γιατί θα το δούμε αυτό να επαναλαμβάνεται ως αντίδραση από το Συμβούλιο, συνεχώς θα μπλοκάρουν και νομίζω ότι όλα τα μέρη εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξουν την πρόταση της κυρίας Ρέντινγκ και πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε επί αυτής της οδηγίας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τρίτη συγγήτρια, κυρία Γιανακουδάκη. Θεωρώ ότι μιλάμε γενικά για την πρόταση αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, πρέπει να αποσαφηνίσω ένα σημείο που δεν ανέφερε η καλή μου φίλη. Ότι έχει διαρρεύσει αυτή η εκθέση. Έτσι λοιπόν δεν ξέρουμε τι ακριβώ περιλαμβάνει, αλλά εργαζόμαστε επί υποθέσεων. Δεν ξέρουμε πώς έχουν προταθεί Η περίοδος διαβούλευσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη για την έκθεση αυτή. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είχε ολοκληρωθεί. Προέτρεχα μάλλον. Λοιπόν, να σα αναφερθώ στο Συμβούλιο τότε. Νομίζω ότι το Συμβούλιο ε, αποτελείται από εκλεγμένους αξιωματούχους, απαραίτητους. Ε, ναι, γιατί έχουν, ε, υπάρχουν μέλη της κυβέρνησής σας στο Συμβούλιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βασίλειο είναι εκεί. Has the floor now, please. Συγχωρείτε κυρία έχει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, Α υποθέσουμε ότι όσοι πηγαίνουν στο Συμβούλιο είναι από τι εκλεγμένε κυβερνήσει, ε, όπω γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζω και εσεί να έχετε εκλεγμένε κυβερνήσει. Δεν ε, καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αντιδρούμε στο Συμβούλιο, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε μαζί του. Και κάτι άλλο. Υποθέτω ότι όλοι πιστεύουμε στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 16 υπάρχει ελευθερία να ε, ιδρυθεί μια επιχείρηση και το άρθρο 21 απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου. Έτσι λοιπόν ε, μπορούμε να εργαστούμε βάσει αυτών, κυρίες μου. Πρόεδρος. Έχουμε μακρύ κατάλογο ατόμων που έχουν ζητήσει το λόγο. Έτσι λοιπόν θα συζητούσα να μην μακρηγορείτε για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να τους ακούσουμε όλους όσους επιθυμούν το λόγο. Ας περάσουμε στην κυρία Καμπριέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα χώριζα σε δύο τμήματα την παρέμβασή μου. Πρώτα απ' όλα για μια ακόμη φορά θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε η συνάδελφός μα η κυρία Κράτσα. Πράγματι περιμέναμε πάρα πολύ μέχρι ότου οι κυβερνήσει και οι εταιρείε να δείξουν κάποια προθυμία και να εφαρμοστούν τα μέτρα που στηρίζουμε για να ισχυθεί η θέση των γυναικών. Υπάρχει αυτή η διαπίστωση. Εμεί συνεχώ αυτό συζητάμε. Αντίθετα όμω, εδώ πρέπει να τεθεί ένα ερώτημα. Ποιο είναι ο στόχο μα, ε, ποιον θέλουμε να πείσουμε, δεν νομίζω ότι αυτή η δουλειά τη πυθού θα πρέπει να γίνει εντό τη Επιτροπή Γυναικών, ούτε εν πάση περιπτώσει αν γίνει εντό Επιτροπή Γυναικών, μετά την περιπτώση υπάρχουν δύο απουσίε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα η Επίτροπο Ρέντινγκ να είναι μαζί μα για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε το θέμα. Ό, όχι την υποστήριξη για την πρωτοβουλία τη, όμω τι λεπτομέρειε τα βήματα τα συγκεκριμένα ούτω ώστε να μεταμορφωθεί η υποστήριξη σε αποτελέσματα. Και δεύτερον, θέλω να υπογραμμίσω ότι ποτέ δεν έχουμε προτάσει συγκεκριμένε. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο καρποφόρο να είχαμε μια βάση πιο στερεή και από πλευρά ατόμων που συζητούν και από πλευρά κειμένου επί το οποίο θα μπορούσαμε να εστιαστούμε. Ε, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω ίσως προσωπική άποψη αυτή Σίγουρα υπάρχουν χώρε που ήδη έκαναν, είχαν κάποιε αντιδράσει. Εγώ θα ήμουν πολύ πιο προσεκτική. Ίσως είναι και ένα από τα αποτελέσματα boomerang τη ΜΜΕΝ που δεν αντιδράσαμε εμεί. Εδώ και ένα χρόνο υποστηρίζαμε μια πρωτοβουλία που δεν ετέθη επί χάρτου ξεκάθαρα, μαύρο σε άσπρο, αλλά από την άλλη θετικό μήνυμα αποδεικνύει ότι ακολουθούμε σωστή κατεύθυνση, είμαστε στο καλό μονοπάτι. Αν χώρες αντιδρούν τόσο μπορούμε και εμείς πραγματικά να βασιστούμε στην υποστήριξη των πολιτών. Διότι εδώ τους πολίτες προστατεύουν στο Κοινοβούλιο και αυτό δείχνει ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε. Εξού και η προσοχή που δίνουμε και πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες ούτως ώστε τα αποτελέσματα τελικά να τα πετύχουμε. Για ακόμη μια φορά αποτελέσματα μόνο όταν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, όταν έχουμε ένα κείμενο, όταν υπάρχει συζήτηση, ένα διάλογο, όχι διάλογο μεταξύ μα, μόνο τότε θα πετύχουμε. Εδώ στην Επιτροπή Γυναικών δείξαμε επανειλημμένα ότι η κυρία Ρέντινγκ μπορεί να στηρίζεται πάνω μα. Θα θέλαμε επίση κάθε βήμα μπροστά να γίνει μέσω διαλόγου και χέρι με χέρι. Εκφράζω ακόμη μια φορά τη λύπη μου που τώρα εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με εκείνη ή με κάποιον που την εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί το γραφείο τη, ώστε αυτή η συζήτηση τελικά πραγματικά να είναι αποτελεσματικότερη, που πιστεύω ότι είναι πρωταρχική σημασία. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Χάνιμπολ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ότι δεν έχουμε κάτι μπροστά μας και ότι συζητούμε το θέμα σήμερα οφείλεται σε δράσεις κάποιων κυβερνήσεων κρατών μελών και μία από αυτές τις χώρες είναι η δική μου και κυβέρνηση και ντρέπομαι πάρα πολύ από τη συμπεριφορά της Βρετανικής κυβερνήσεως σε αυτή την περίσταση και θέλω να καταχωρηθεί αυτό. Δεν το συνηθίζουμε στην Επιτροπή αυτή ούτε στο Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εκτελήσονται τα πράγματα υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να κατηγορηθούν για την εξέλιξη και αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε θα ήταν να τα διορθώσουμε από τα πράγματα. Εγώ πάντα υποστήριζα ένθερμα την πρωτοβουλία της κυρίας Ρέντινγκ. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εκπροσωπούνται στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών οι γυναίκες σε όλη την Ευρώπη, στι περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στον Ηνωμένο Βασίλειο, είναι κάτι απέσιο, φρικτό. Λιγότερο από 10% των θέσεων υψηλών στελεχών στις εταιρείε κατέχονται από γυναίκες και νομίζω ότι είναι και η ώρα να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και ο τρόπο με τον οποίο το προσήγγιζε η κυρία Ρέντινγκ ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν επεβάλλωτο. Επέρναγε από διαβουλεύσει. Και είναι κρίμα, πραγματική τραγωδία είναι, ότι καταλήγει με αυτόν τον τρόπο. Που τελικά δείχνει να διαμορφώνεται σε ε, χάλι, ε, σε μια φάρσα. Δεν θα πρέπει να χάσουμε το θέμα. Σαν μέλη τη Επιτροπή πρέπει να πούμε στην κυρία Ρέντινγκ ότι την υποστηρίζουμε πάρα πολύ να έρθει εδώ να τις μιλήσουμε για το θέμα και σαν Επιτροπή Γυναικών και Κοινοβούλιο να είμαστε ενωμένοι διότι είμαι σίγουρο ότι θα περάσει από την Ολομέλεια όταν στρωθούμε. Υπάρχει ομοφωνία στις ομάδες, εκτός από μια αξιοσημείωτη εξαίρεση που αναμέναμε. Έχω την πεποίθηση λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει με αυτό. Άρα θα είναι θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κατά του Συμβουλίου. Κλασική περίπτωση. Και ούτε ε, θα έχουμε την πλειοψηφία του Συμβουλίου, θα έχουμε ε, την μπλοκάρουσα μειοψηφία. Απορτίζεται από εκλεγμένες κυβερνήσεις κρατών μελών το Συμβούλιο, αλλά δεν δρούν τι ούτω τρόπος. Και λίγες χώρες, εννέα από ό,τι ξέρω από τις μυστικές πληροφορίες που έχω, εννέα χώρες στο Συμβούλιο θα αντιταχθούν δεν είναι η πλειοψηφία. Και θα είμαστε πιθανότατα στη θέση όπου θα έχουμε την πλειοψηφία των επιτρόπων, την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και θα κολλήσει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Και τι πράγματι συζητάμε. Συζητάμε ένα μέτρο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη διάκριση και τα βασικά δικαιώματα, να δώσουμε στις γυναίκες την εκπροσώπηση που θα έπρεπε να έχουν και πέραν αυτού, σαν αποτέλεσμα αυτό που είπε και η κυρία Κράτσα, έχει γίνει έρευνα που δείχνει ότι οι εταιρείε τα πηγαίνουν καλύτερα όταν έχουν καλύτερο μείγμα, περισσότερε γυναίκε στα διοικητικά του συμβούλια. Λοιπόν, αυτό που κάνει μπλοκάρισμα με ψηφία στο Συμβούλιο είναι φρικτό. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθούμε απέναντί του και να είμαστε σίγουροι ότι στο τέλο τελικά το μέτρο θα γίνει αποδεκτό. Ε, κυρία Η ομάδα μας, η ομάδα των Πρασίνων, έστειλε μία επιστολή στον κύριο Μπαρόσο για να υποστηρίξει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ζητήσει να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν μία διαδικασία νομοθετική. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει επουδενή να υποχωρήσουμε σε πιέσεις οι οποίες είναι σκανδαλώδεις και η διαδικασία λήψη αποφάσεων η Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιριών είναι γελία χαμηλά συμφωνούμε όλοι πάνω σε αυτό, και ο αριθμός των ε, γυναικών που είναι ικανές δεν είναι πολύ μικρός, αντίθετα από αυτά που σκέφτονται κάποιοι. Ε, μπορούμε να δούμε ότι οι γυναίκες ειδικευμένες είναι πάρα πολλές. Το 2010 οι γυναίκες ήταν το 60% των διπλωματούχων με δίπλωμα πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα, δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε σε αυτές τις πιέσεις τις οπισθοδρομικές, θα πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα. Ähm, Κυρία ähm, Ευχαριστώ. Και οι φιλελεύθεροι υποδέχονται θετικά την πρόταση της Επιτρόπου Ρέντι. Είμαστε ικανοποιημένοι που θα ξεκινήσει αυτή η νομοθετική διαδικασία και δεν ε, θέλουμε να βασιζόμαστε μόνο σε ελπίδες και υποθέσεις για το μέλλον αλλά θα θέλαμε να περάσει σε επίσημους διάβλους, ε, σε διάφορα κρατημέλη. Αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν ορισμένα κρατημέλη τα οποία έχουν εισαγάγει μια ιδιαίτερα φιλόδοξη νομοθεσία που πηγαίνει πολύ παραπέρα και δεν ε, αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, και σε ό,τι αφορά τις ε, ποσοστώσεις για τις γυναίκες και οι προτάσεις ε, ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη και νομοθεσία, όπως σας είπα, είναι πολύ πιο φιλόδοξη. όπως είπε και η κυρία Κράτσα, θα πρέπει να κατανοήσουμε ποιος ε, έχει φωνή στο θέμα αυτό στην Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν ε, για έναν διαγωνισμό μεταξύ των ε, διάφορων θεσμών, μεταξύ των διάφορων οργάνων. Η Κομισιόν κανονικά παρουσιάζει τις νομοθετικές προτάσεις, όμως πολλές φορές έχουμε αντιδράσει από το Συμβούλιο, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μπορώ να σας πω ότι ήταν ουσιαστικά και κάπως συναισθηματικού χαρακτήρα οι αντιδράσεις. Ε, όλα αυτά ε, δεν αρμόζουν σε μια νομοθετική πρόταση, όμως ε, μπορώ να σας πω ότι... ο Γερμανός αντικαγκελάριος δεν εκλέγεται από τους πολίτες, αλλά διορίζεται από τη Γερμανίδα καγκελάριο. Κατόπιν ε, υπάρχουν ε, και διαφορετικές δημοκρατικές διαδικασίες ε, σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους στο Συμβούλιο. Ενώ εμείς εδώ εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν ε, είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να αποφύγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα λάβει υπόψη όλα αυτά, γιατί έχουμε διάφορους υπουργούς και υπουργοί που είναι εντελώς αντίθετοι. Όμως υπάρχουν άλλοι που είναι θετικοί στην πρόταση της κυρίας Ρέντινγκ. Έτσι λοιπόν, ακόμη και στο εσωτερικό της Γερμανίας δεν είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι, ότι είναι όλοι εντελώς αντίθετοι. Εξαρτάται από το ποιος θα καθίσει στην ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν, αυτή η κατάσταση δείχνει ποια είναι η θέση μας. Να σας πω ότι η Επίτροπος ε, Ρέντινγκ ήταν πολύ αποφασισμένη και θέλει να κάνει κάποια βήματα προς τα μπρος, να προωθήσει κάποιες προτάσεις και... Τελικά, βέβαια δεν υπήρξαν ε, στην πραγματικότητα πολύ μεγάλα αποτελέσματα, υπήρξαν μακρές διαβουλεύσεις μέχρι το Μάιο, τώρα στο το φθινόπωρο θα έχουμε μία πρόταση και φυσικά θα πρέπει να περάσει από όλε τι γενικέ διευθύνσει ε, για να τοποθετηθούν και οι γενικέ διευθύνσει, να γνωμοδοτήσουν και κατόπιν θα περάσει από το Σώμα των Επιτρόπων. Πάντα το φθινόπωρο. Και πρέπει να σας πω ότι στο εσωτερικό της Κομισιόν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, κυρίως ε, από αυτούς ε, που έχουν φτάσει να κατακτούν κάποιες θέσεις σε βάση ποσοστώσεων. Υπάρχει διαφορά όταν μιλούν κάποιες για τον εαυτό τους ή μιλούν για την ισότητα των δύο φύλων σε ορισμένα πλαίσια οικονομικά. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα έπρεπε να πράξουμε κάθε τι δυνατόν, να βάλουμε τη δυνατά μας ε, για να δώσουμε συνέχεια στα όσα κάναμε μέχρι τώρα και εμείς ε, ως ε, φιλελεύθεροι γράψαμε και στον κύριο Μπαρόσο με επιστολή βέβαια δεν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης και νομίζω ότι είναι κρίμα γιατί θα μπορούσε να ε, δείξει σε εκείνη την περίπτωση για μια ακόμη φορά ότι λαμβάνει σοβαρά ο πρόεδρος της Κομισιόν να συζητούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να δείξουμε εμεί ως Επιτροπή ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξη της κυρίας Ρέντινγκ προκειμένου να δείξουμε ότι εμείς συνεχίζουμε με τόσα κάναμε στο παρελθόν στις ψηφορίες μας. Επόμενο μιλήτρια, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λέει κυρία Λούνατσεκ. Συμφωνώ με όσου είπαν ότι υποστήριξε, πρέπει να υπάρξει σοβαρή υποστήριξη από τη δική μα επιτροπή στην Επίτροπο Ρέντινγκ για να προχωρήσει με την πρότασή τη. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα, στο περιεχόμενο και στη διαδικασία. Ω προ το περιεχόμενο, όπω είπαν και πολλοί Άλλοι υπήρξαν πολλές ε, αποδείξεις, έχουν υπάρξει αποδείξεις ότι αν ε, υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση στα συμβούλια και από τα δύο φύλλα, τότε οι εταιρείε θα πάνε καλύτερα. Και θέλω να υπενθυμίσω όσους, ε, ήταν επικριτικοί στην πρόθεση της κυρίας Ρέντινγκ. Ε, πριν ένα, ένα μισή χρόνιο είπε η κυρία Ρέντινγκ, ώρα θα ζητήσω από όλου ε, να το κάνουν εθελοντικά. Αλλά δεν έκαναν όσα πρέπει και τότε είπε ότι αν δεν λειτουργεί ο θελοντισμό, τότε θα πρέπει να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Και εγώ νομίζω ότι είναι φυσικό. Αν ε, δεν λειτουργούν τα πράγματα σε κούσια βάση, και επίση ε, και μια μεγάλη γκάμα επιστημόνων ε, πιστεύουν και είναι αποδεικμένο αυτό ότι είναι καλό να έχουμε ε, ισότιμη εκπροσώπηση, τότε θα πρέπει να έχουμε υποχρεωτικό χαρακτήρα και η επιστολή των νέων υπουργών του Συμβουλίου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λένε ότι είναι υπέρ να εκπροσωπούνται ισότιμα και οι γυναίκες, αλλά κατόπιν αναφέρονται στην αρχή της επικουρικότητας και λένε ότι πρέπει να το κάνουν. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει εδώ και ένα μισή χρόνο από τότε που το ανέφερε πρώτη φορά η κυρία Ρέντινγκ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι λογικό η κυρία Ρέντινγκ να προχωρήσει τώρα και εμεί να την υποστηρίξουμε. Αυτό επί του περιεχομένου. Τώρα, σχετικά με τη διαδικασία. Υποστηρίζω την πρόθεση να γράψει δική μας, να συντάξει μια επιστολή δική μας επιτροπή Προ τον πρόεδρο Μπαρόζο, αλλά ίσω και προ το Συμβούλιο. Προκειμένου να δηλώσουμε πόσο πολύ διαφωνούμε με τα μέλη του Συμβουλίου, είτε είναι εκλεγμένα είτε όχι. Δεν εκλέγονται ούτε στη δική μου χώρα. Δηλαδή εκλέγεται το Κοινοβούλιο και κατόπιν ε, βάσει πλειοψηφία ε, σχηματίζεται την εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση. Έχουμε διαφορετικέ μεθόδου λοιπόν, ε, το πώ ε, συστήνεται η κυβέρνηση στα διαφορετικά μέλη, αλλά τέλο πάντων. Και θα πρότεινα λοιπόν εμείς από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών να ζητήσουμε από την Προεδρία αυτού του Κοινοβουλίου επίσης να απευθυνθεί στο Συμβούλιο σε σχέση με τη διαδικασία όπως είπαν και άλλοι προκειμένου και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι αντιπρόεδροι να απευθυνθούν στο Συμβούλιο και να του πούν «Κοιτάξτε, πρόκειται για μια διαδικασία εδώ που αντικείται στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική διαδικασία. Α μην το κάνουμε εμεί μόνο από τη δική μα Επιτροπή. Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αυτό το θέμα, αφορά την νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Έτσι λοιπόν εγώ θα συνιστούσα από το Προεδρείο τη Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών ή θέλετε να το κάνετε και εσείς ο ίδιο αν θέλετε Πρόεδρε να ζητήσετε από την Προεδρία να στείλει μια επιστολή στο Συμβούλιο και να τους πει δεν είναι σωστός τρόπος να αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Και κάτι άλλο, ε, κυρία Ιεράνα, άκουσα σωστά. Αναφερθήκατε σε επιτρόπους που υποτίθεται ότι είπαν ότι είναι κατά. Ναι, το ξέρω η Αντιπρόεδρος Άστον και η επίτροπο Μάλστρομ ήταν κατά την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Κάποιε από εμά απευθύνθηκαν σε αυτέ προσωπικά και μα είπαν ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Ίσως ε, να μην είναι ισχυρέ υποστηρίκτριε, ίσω θα προτιμούσαν να μην χρειάζονται ποσοστώσει, αλλά δημοσίω είπαν ότι όχι. Δηλαδή υπήρξε κάποια σημαίνει πληροφορία και νομίζω ότι ήταν καλό να το πολυθεύσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλου τρει συναδέλφου που έχουν συζητήσει το λόγο και κατόπιν θα ακούσουμε του εκπροσώπου τη Κομισιόν και του Συμβουλίου ίσω και να δούμε αν θα έχουμε και χρόνο για άλλε παρεμβάσει. Αλλά καταρχήν α ακούσουμε ποιον δεν έχει μιλήσει ακόμα και να δούμε και αν εκπρόσωποι από το Συμβούλιο και την Επιτροπή θέλουν να πούν κάτι ακόμη. Παρακαλώ, κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σκέψεις πολύ σύντομες. Οι γυναίκες ε, στην Ευρώπη ε, αποτελούν το 60% ε, όσων έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, έχουν προσόντα και έχουν ε, τι ικανότητε για να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Τι συμβαίνει, ότι στην πραγματικότητα ε, υπάρχουν κάποιες περιστάσει που τους ξεπερνούν. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία της κυρίας Ρέντινγκ. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ακολουθεί την έκκληση και την πρόσκληση των κρατών μελών για αυτορύθμιση με μια αποδεκτή χρονική περίοδο έτσι ώστε να κάνουν οι χώρες αυτή την αυτορύθμιση. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έγινε και επομένως είναι απόλυτα λογικό η Αντιπρόεδρος τώρα να παρουσιάζει μια νομοθετική πρόταση έτσι ώστε το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τη σχετική νομοθεσία και να θέσουν σε εφαρμογή την νομοθεσία αυτή για να τεθεί αυτό το θέμα της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων. Θα πρέπει το Κοινοβουλίο να δώσει πολύ σαφή μηνύματα ότι υποστηρίζει την πρόταση της Αντιπροέδρου και θα πρέπει, όπως σας είπα, να δώσει αυτό το μήνυμα και εγώ εδώ ε, ουσιαστικά μιλώ εκ μέρους μιας χώρας που βιώνει μια πολύ σοβαρή κρίση οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική. Αυτή η σοβαρή κρίση δεν μπορεί να αποτελεί πρόφαση για κανένα μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να μην συνεχιστεί αυτή η κατάκτηση των ίσων δικαιωμάτων μεταξύ των δύο φύλων. Και είναι ουσιαστικό να μην ε, χρησιμεύσει αυτή η μεγάλη κρίση ως πρόφαση σε αυτόν τον αγώνα για την κατάκτηση των δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συντονισμό με την ε, Αντιπρόεδρο, την κυρία Ρέντινγκ, να δώσει τα κατάλληλα μηνύματα και να λάβει τις απαραίτητες σαφείς πρωτοβουλίες για να δείξει ότι εμείς ε, δεν συμφωνούμε με αυτή την εμπλοκή που γίνεται αυτή τη στιγμή και μάλιστα χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί επισήμως η πρόταση και χωρίς να έχει μπει στην ε, νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι σε αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, αφορά τον πολιτισμό μας και αφορά την δικαιοσύνη και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρακαλώ, κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε εκτενώς ε, για αυτές τις περίεργες διαδικασίες και εγώ πιστεύω ότι είναι μια περίεργη διαδικασία αυτή τώρα και το Κοινοβούλιο και η ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλέκονται ε, σε ένα σύστημα το οποίο υπάρχει σχετικά με τις πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει μονοπόλιο των πρωτοβουλειών, άρα η Επιτροπή είναι αυτή η οποία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να το πράξει. Εάν έχουμε κάποιο κείμενο μπροστά μας, βεβαίως τότε θα καταρτήσουμε μία έκθεση σχετικά με αυτό το κείμενο. Εν γνώση μου δεν υπάρχει κείμενο και ε, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί διότι εάν ξεκινήσει ένα προηγούμενο και αρχίσουμε να εμπλεκόμαστε σε μία ιδέα κάποιου επιτρόπου ο οποίος σκοπεύει να αναλάβει μία πρωτοβουλία τότε αλλήμονό μας. Ο κάθε επίτροπος τότε θα πρέπει να ε, στρέφονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν καν ε, απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από φόβο ε, του να μην επιτύχουν πλειοψηφία. Αλλά γνωρίζω την κυρία Ρέντινγκ γιατί ήμουν συμμαθήτρια με τη μητέρα της στο γυμνάσιο και νομίζω ότι είναι απολύτως σε θέση να πείσει η κυρία Ρέντινγκ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Επιτροπή εξαρτάται και όχι από το Συμβούλιο. Όταν λοιπόν αντιδρά η Επιτροπή, ίσως αντιδρά διότι ακριβώς υπάρχει αυτή η ιδιόμορφη διαδικασία όπου προσπαθούμε να προκαταλάβουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το μονοπόλιο των πρωτοβουλειών της, δηλαδή ε, ε, υπέρ ε, της διαδικασίας αυτής και επειδή είναι για καλό σκοπό, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο κοινοβούλιο που μάχονται για την ισότητα των ευκαιριών των γυναικών όσο εγώ δεν νομίζω ότι ε, καμία άλλη δεν ξεκίνησε την ε, δεκαετία του 60 και ορισμένες δεν είχαν καν γεννηθεί. Οπότε δεν θέλω να μου κάνει κανείς μαθήματα, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αναλαμβάνει κανείς ε, δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να είναι ε, ε, αντιπαραγωγικές για τις ε, γυναίκες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υποβάλουμε τις προτάσεις μας ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του μονοπωλίου των πρωτοβουλειών της να μας διατυπώσει προτάσεις τις οποίες στη συνέχεια μπορούμε να αναλύσουμε και αναλόγως εάν είναι καλές ή αν τις τροποποιήσουμε και τις φέρουμε στα μέτρα μας να τις ψηφίσουμε ε, θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή για αυτή την ιδιόμορφη διαδικασία η οποία εφαρμόζεται για να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω σε ποιον. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Ο κύριος Μπαρόζο ξέρει τι θέλουμε. Έχουμε υιοθετήσει πάμπολα ψηφίσματα και εκθέσεις όπου λέμε σαφώς και ρητός τι θέλουμε. Τώρα το να στηρίξουμε, ε, μη, να βασιστούμε σε μία πρόταση κάποιου επιτρόπου που ακόμη δεν έχει οθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω ότι ε, το προηγούμενο αυτό είναι ιδιόμορφο και δεν θα ήθελα άλλοι επίτροποι, ιδίως αν έχουν ε, περίεργες ιδέες, να έρχονται οι επίτροποι αυτοί στο Κοινοβούλιο, να κάνουν μία εκστρατεία για να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προωθήσουν ίσονες ιδέες τις οποίες δεν συμμερίζονται οι ομόλογοι τους. Διότι αν τις συμμεριζόντουσαν γιατί δεν θα προχωρούσαν. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στη διαδικασία αυτή την οποία έχετε υιοθετήσει και η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήταν πολύ κακή υπηρεσία σε μια πρωτοβουλία που οι περισσότεροι από εμά συμμερίζονται εάν προχωρούσαμε και γράφαμε ε, μια επιστολή εν ονόματι μιας πλειοψηφίας που δεν εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο. Εάν δούμε ότι η πρόταση της κυρίας Ρέντινγκ δεν περάσει, δεν υιοθετηθεί δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα πρέπει να επέμβουμε, όχι όμως τώρα. Τώρα πρέπει να αφήσουμε το μονοπόλιο της πρωτοβουλίες και τις ευθύνες σε όλους τους επιτρόπους για να πούν εάν υιοθετούν μια τέτοια πρόταση ή όχι. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπέρμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μπορώ να συμφωνήσω με ποτέ, ε, πολλές προτάσεις οι οποίες έγιναν συγκεκριμένα για την στιγμή. Ε, είδαμε από την κρίση ότι οι γυναίκες στις βασικές στις, στις βασικές αποφάσεις εάν είχαν συμμετάσχει στη λήψη τους γυναίκες δεν θα υπήρχε κρίση. Άρα είναι πολύ πιο βασικό τώρα να αυξηθεί η ποσόστοση των γυναικών από ό,τι στο παρελθόν ή από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Θεωρώ ε, δε ότι είναι ε, μία, ένα πλήγμα προς τη δημοκρατία και οι γυναίκες είναι μέρος της δημοκρατίας και άρα πρέπει και εμείς ε, να συμμετέχουμε στο μέτωπο για να μπορούμε όλοι μαζί να μπορέσουμε να εκφράσουμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας, διότι ε, ε, θα ήθελα να στηρίξω την πρόταση της ε, συναδέλφου Λούνα Τσεκ νομίζω ότι είναι πολύ σωστή πρόταση για να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ε, εάν θέλει να λάβει τον λόγο και αν θέλει για πολύ σύντομα γιατί ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η Επιτροπή. Το όνομά μου είναι Ντανιέλα Μπανκιέ, είμαι ε, η επικεφαλής ε, της, ε, του τομέα της α, ε, και συνεργάζομαι με την Κενήρια Ρέντινγκ εναντίον των διακρίσεων. Άκουσα τη συζήτησή σας και τις αντιδράσεις σας. Ήθελα λοιπόν να πω ουσιαστικά ένα πράγμα και αυτό είναι ότι η ιδέα του να προτείνει κανείς ένα μέτρο για να προωθηθούν οι γυναίκες στην οικονομική ηγεσία δεν ε, είναι έκπληξη και δεν ήταν ε, ποτέ ε, μυστικό ούτε κανείς έχει αποκρύψει τίποτα. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2010 και ε, είναι μία ε, απόδειξη μία στρατηγικής μεταξύ ανδρών και γυναικών όπου προωθούνται πέντε πρωτοβουλ... Ε, προτεραιότητες και το 2011 υπήρχε μία δέσμευση της Επιτροπής προς τις επιχειρήσεις ότι οι επιχειρήσεις οικειοθελώς θα δεσμεύσουν έναν αριθμό θέσεων για γυναίκες στα συμβούλια των ε, επιχειρήσεων που θα είναι 15% ε, αρχικά και 20% μέχρι το 2020. Στη συνέχεια η Επιτροπή προώθησε τις προσπάθειες αυτές της αυτορυθμίσεως των επιχειρήσεων το 2012 και αναφέραμε τους πρόσφατους αριθμούς σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στα συμβούλια των επιχειρήσεων επιχειρήσεων ε, δημοσιεύθηκε στην έκθεση του Μαρτίου και η Αντιπρόεδρος προέβη σε μία δημόσια διαβούλευση για τα καλύτερα μέτρα για να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στα Συμβούλια των Επιχειρήσεων και πρότεινε να υπάρξει και αργότερα μία πρωτοβουλία η οποία αναφέρεται και στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σύντομα μία διευκρίνηση σχετικά με την διαδικασία που έχουμε αυτή τη στιγμή γιατί υπήρξαν ορισμένα ερωτήματα. Ισχύει ότι η πρόταση της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ συζητείται μεταξύ των υπηρεσιών, δηλαδή είναι στο τεχνικό επίπεδο για σχόλια μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, συνεχίζεται και όταν, και θα, θα ολοκληρωθεί θα συζητηθεί σε επίπεδο επιτρόπων. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποια στιγμή θα υιοθετηθεί και έχουμε δει πόσο ενδιαφέρουσα είναι η συζήτηση και ε, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει στο πρόγραμμα εργασίας ότι θα υιοθετηθεί η πρόταση πριν το τέλος του έτους. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ε, περιεχόμενο της προτάσεως, σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Όταν θα υπάρξουν τα στοιχεία και η κυρία Ρέντινγκ και οι υπόλοιποι θα θελήσουν ε, να συζητήσουν λεπτομέρειες. Προς το παρόν υπάρχουν αυτά που διαβάσατε στον τύπο. Δηλαδή ότι το βασικό χαρακτηριστικό της προτάσεως ε, ε, αναφέρεται στις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και οι οποίες πρέπει να διαθέσουν 40% 10% θέσεων σαν στόχο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, οι εταιρείες του κράτους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, ε, όλες αυτές περιλαμβάνονται. Άπαξ λοιπόν και μια τέτοια πρόταση διαρρεύσης στον τύπο ε, λαμβάνεται, κατακλείζεστε μάλλον από επιστολές και η κυρία Ρέντινγκ όπως και όλοι οι άλλοι επίτροποι γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του γενικώ ότι δεν υπάρχει ε, μία μειοψηφία που μπορεί να μπλοκάρει την πρόταση της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό μπορεί να γίνει κάπως αργότερα αλλά και επαναλαμβάνω με αυτή τη στιγμή η κυρία Ρέντινγκ θεωρεί ότι πρέπει πρώτα η διαδικασία να κινηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά να υποβληθεί στους συνομοθέτες και αυτοί θα αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, στην διαδικασία. Το άλλο που ήθελα να σας πω, διότι υπήρξαν ορισμένες παρατηρήσεις για την οικονομική σημασία και για τη διάσταση των βασικών δικαιωμάτων, είναι ότι υπάρχουν ε, αξιολογήσεις των επιπτώσεων που θα συνοδεύσουν την ε, πρόταση. Έχουμε εξετάσει επιπτώσεις και στο ε, μικροοικονομικό επίπεδο για τις επιχειρήσεις και στο μακροοικονομικό για την οικονομία των κρατών και είναι ένα στοιχείο πυρήνας στην πρόταση Επιπλέον βασιζόμαστε στον χάρτη των βασικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η διάκριση βάση του φύλου και θέλω να πω πολύ σύντομα ότι βεβαίως έχουμε εξετάσει λεπτομερέστερα την εμπλοκή του χάρτη των βασικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας διεκπαιρεώσεως εργασιών και επιχειρήσεων. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει αναλογικότης και να υπάρχει μία εξήγηση για τους περιορισμούς. Δεν είναι απεριόριστα όλα και ο χάρτης των βασικών δικαιωμάτων ο, ε, δηλαδή, τόσο αναφέρει ότι δεδομένων δράσεων, ορισμένων δράσεων πρέπει να δίδονται ε, και να επιτρέπεται να δίδονται ορισμένα ωφέλη σε μέρη του πληθυσμού και πρέπει και από αυτή την οπτική γωνία να κοιτάξουμε το θέμα. Τώρα θα ρωτήσω εάν ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου θέλει να σχολιάσει, πράγμα που δεν είναι υποχρεωτικό, τότε επειδή έχουμε πέντε μόνο λεπτά θα ήθελα κυρία Κράτσα να ολοκληρώσει. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι ομιλητές στον κατάλογο, αλλά είναι δυνατόν και αυτοί ενδεχομένως να πούνε μια κουβέντα. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω τώρα, εάν η κυρία Μορβάη έχει κάτι ακόμη να πει, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Κράτσα. Επιτρέπετε κυρία Κράτσα ε, για πολύ σύντομο διάστημα. Ευχαριστώ. Ο, κατάλαβα αυτό που είπε η Επιτροπή να περιμένουμε μέχρι ότου καταρτιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Στην περίπτωση όμως αυτή, γιατί υπάρχουν ήδη νέα κυβερνήσεις ε, εκδηλώθηκαν και είπαν ότι δεν θέλουμε αυτή την πρόταση. Ε, η δικιά μου κυβέρνηση που συγκαταλέγεται στις εννέα κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη, ε, κάτι έχω στο νου τους και θέλουν να προστατεύσουν την ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν θέλουν αλλαγές και ε, εξέφρασαν τις απόψεις τους. Είπαν ότι δεν θέλουν την πρόταση αυτή. Οπότε εμείς ε, ε, δεν πρέπει να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Είμαστε εδώ γυναίκες και άνδρες που είμαστε πολιτικοί, που θέλουμε αλλαγή, που θέλουμε να αλλάξουμε την ισχύουσα κατάσταση και αν αυτοί ε, προστατεύοντας την ισχύουσα κατάσταση έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους γιατί και εμείς να μην έχουμε την ίδια δυνατότητα και την ίδια ελευθερία. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα τον τελευταίο λόγο στην κυρία Κράτσα πάρα πολύ. Εγώ είμαι βιαστική, έχω ένα ραντεβού ήδη στις 6 και 4. Ε, λοιπόν, καταρχάς να διευκρινίσω τη δική μου θέση. Εμένα η δική μου θέση δεν είναι ότι πρέπει να παρέμβουμε στη διαδικασία την νομοθετική. Εγώ έχω κάνει ερώτηση στον κοινοβουλευτικό μας έλεγχο ήδη τον Ιούλιο και έστειλα και επιστολή στον πρόεδρο στον κύριο Μπαρόζο. Η επιστολή μου, το περιεχόμενο της παρέμβασής μου δεν έχει να κάνει με το να του υποδεικνύουμε τι πρέπει να κάνει ως πρόεδρος Επιτροπής. Είναι βασισμένη στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνόδευσε την έκθεσή μου, που λέει ότι δίνουμε περιθώριο ένα χρόνο στην Επιτροπή, εάν δεν υπάρχει εξέλιξη και οθελής στην συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, να φέρει νομοθετική πρόταση. Τον Ιούλιο λοιπόν ρωτάω, ζητά, κούρω ε, τον κόδωνα του κινδύνου και λέω πέρασε ο χρόνος που σας είχαμε δώσει περιθώριο. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Και στον κύριο Μπαρόζο επανήλθα, αν δεν είχε δημιουργηθεί αυτό, αυτό το θέμα, για να είμαι ειλικρινής δεν θα έγραφα στον κύριο Μπαρόζο, θα έμενα στην ερώτηση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έγραψα όμως βασισμένη όχι στους θορύβους, στο να του απαιτώ για ένα σημαντικό θέμα που το, που το αιτιολόγησα ότι είναι σημαντικό, να δώσει απάντηση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι εκεί θα εμείς να παρέμβουμε σε ό,τι έχει να κάνει με, το, με τη δική μας θέση και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της το ψήφισμα του 11 που έλεγε ότι μέχρι τον Ιούλιο του 12 πρέπει να φέρει νομοθετική πρόταση. Και έτσι έμεσα βοηθάμε βέβαια την υπόθεση. Όταν είπα να αντιδράσουμε στην κοινή γνώμη, ενώ ως πολιτική, όπως λέει η κυρία Μορβάη, που μας ρωτούν διάφοροι δημοσιογράφοι, βουλευτές από τη χώρα μας, τι γίνεται με μια πρόταση που βρίσκεται. Εκεί εμείς ως πολιτικοί και ως φορείς αυτής της ιδέας για το Κοινοβούλιο έφερε από πέρυσι αυτή την ιδέα, πρέπει να, δημιουργεί, να φτιάξουμε αντισώματα στη κοινή γνώμη και να εξηγούμε όταν μας ρωτούν τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση. Ότι είναι κάτι που το Κοινοβούλιο το έχει ψηφίσει, το στηρίζει, ε, ήταν πρόδρομος και άνοιξε το δρόμο και στην κυρία Ρέντινγκ, γιατί η κυρία Ρέντινγκ ήταν πολύ ευτυχής με το ψήφισμά μας, διότι ήταν για αυτήν ένα όπλο να μπορέσει να περάσει την πρόταση. Αισθάνομαι ότι έχουμε όλα τα επιχειρήματα στο Κοινοβούλιο να ε, δημιουργήσουμε μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα χωρίς να παρέμβουμε στη δουλειά που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε πρέπει να φύγω. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα απλώς να κλείσω λέγοντας ότι μόλις θα λάβουμε την πρόταση θα μπορεί να δράσει η Επιτροπή για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να στραφώ και στους συντονιστές και να ρωτήσω πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον, πώς θα μπορούσαμε ίσως να αναλάβουμε δράση πριν από την, πρόταση, πριν από την παρουσίαση της πρότασης. Θα ήθελα οι συντονιστές να πάρουν μία απόφαση σχετικά με το ζήτημα αυτό. Έτσι λοιπόν παρακαλώ να έρθετε και εσείς σε επαφή με τους δικούς σας συντονιστές γιατί είναι σημαντικό και εγώ θα μιλήσω με τους συντονιστές και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την έκθεση της κυρίας Κράτσα σε σχέση με τις ποσοστώσεις που πρέπει να υπάρχουν για τα διοικητικά συμβούλια. Είναι ξεκάθαρη, όπως σας είπα, η θέση του Κοινοβουλίου. Υπάρχει ευρία πλειοψηφία στο ιστορικό του Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. Πριν να κλείσω, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι αύριο θα συνεχίσουμε με ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοκογενειακής βίας κατά των γυναικών. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο ιστορικό αυτή τη επιτροπή, που ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών. Και εδώ ολοκληρώνουμε τη συνεδρίαση και ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από του διερμηνεί, λέει ο πρόεδρο, γιατί καθυστερήσαμε κάποια λεπτά. Σα ευχαριστώ όλους και θα τα ξαναπούμε αύριο.